Good afternoon. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που σας βλέπω. Εδώ ξεκινάμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Πρώτο θέμα, έγκριση της ημερησίας διάταξης. Θα μπορούσαμε παρακαλώ να την εγκρίνουμε. Μάλιστα, περνάμε στις ανακοινώσεις της Προέδρου. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν όλες οι γλώσσες με εξαίρεση τη γλώσσα της Κροατίας, της Φιλανδίας και της Μάλτας. Δεύτερη ανακοίνωση, έκθεση της αντιπροσωπείας έμπλη από τη Βιέννη που έγινε το Μάιο του 2018. Η... Τα στοιχεία θα μπορούσατε να τα βρείτε στα έγγραφα της συνεδρίασης Πρώτο σημείο, η οδηγία για την οποία η είναι η κυρία Κάφταν. Η πρώτη συζήτηση έγινε στο Στρασβούργο στις 12 Σεπτεμβρίου μετά την ε, Ολομέλη και σε μια ιδιαίτερα επικοδομητική ατμόσφαιρα. Παρόλη την ε, εντολή που, τις εντολές που και οι δύο συνομοθέτες εξέφραζαν την επιδημία τους να συνεργαστούν στο μέτρο του Ιδρανικού για να επιτύχουν ένα συμβιβασμό το οποίο θα καταστηστούσε τις ζωές εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών πολύ καλύτερη από τη στιγμή που είναι ο προγωνιαίος λήθος του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Επόμενη συνάντηση στον Οκτώβριο μπορούμε να περάσουμε στο τρίτο σημείο έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 6 Σεπτεμβρίου 2018 δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Από ό,τι βλέπω, εγκρίνεται. Και θα μπορούσαμε να περάσουμε στο σχέδιο γνωμοδότησης. Θα πρέπει να περιμένουμε όμως λίγο για τον εισηγητή. Την κυρία Ιονγκερίος. Επιτρέψτε μου να σταματήσω για λίγα λεπτά και θα συνεχίσουμε.

So, we'll continue. Καλώς ορίσατε και πάλι. Κοινέ διατάξει, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάστο, το Ταμείο Συνοχή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλία και δημοσιονομικοί κανόνε για τα ταμεία αυτά, για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάθεση, το Ταμείο Εσωτερική ασφάλεια και το Μέσο Διαχείριση των Συνόρων και τη Θεωρήση. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία Γιουγκέριο, στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να με περιμένετε. Έκανα έλεγχο στο κτίριο να δω αν υπάρχει προσβασιμότητα για τους ανάπηρους. Μου χρειάστηκε κάποιος χρόνος βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ε, ευκαιρία να εκφράσω τη σκέψη μου σχετικά με τις κοινέ αυτές διατάξεις και τον κανονισμό. Πιστεύω ότι είναι αρκετά κοινό να μιλάμε εδώ για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και εγώ ίδια τη χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή πολύ συχνά. Και βεβαίω είναι λογικό γιατί η αλληλεγγύη αποτελεί μία από τις βασικές αρχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, άρα και που όμως αναργοστιόμαστε τι σημαίνει η αλληλεγγύη στις μέρες μας. Ε, με άλλα λόγια, πώς οι ευρωπαϊκοί λαοί αντιλαμβάνονται στις μέρες μας την αλληλεγγύη. Κατά την άποψή μου, τα επτά ταμεία το κοινό κανονισμό που διαβάσατε ευτυχώ εσείς είναι τα επτά ταμεία που αποτελούν ένα σύμβολο της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Είναι μια έκφραση της κοινή μας επιθυμίας να αναβαθμίσουμε την κοινωνική και οικονομική σύγκληση. Και πραγματικά με χαροποιεί ιδιαίτερα η πρόταση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί μπορεί να μας βοηθήσει να ενδυναμώσουμε την αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση περιορίζει τον κατακαιρματισμό και αυξάνει την ευελιξία και συμβάλλω, είμαι σίγουρη ότι θα συμβάλλει σε μια καλύτερη πρόσβαση στα ταμεία, πράγμα που σημαίνει ότι τα τελικά περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν άμεσα να ωφεληθούν από αυτά τα ταμεία. Παρ' όλα αυτά, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Το 2014 ο πρόεδρος Ιούνκερ ε, πρόσθεσε το τριπλό α και με την δήλωση του έθεσε τα κοινωνικά θέματα ακόμα πιο ψηλά στο χρονοδιάγραμμα της Ευρώπης. Δυστυχώς το ευρωπαϊκό πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που, που έκυψε από αυτό το τριπλό α δεν αναφέρεται εκτενώς στο, στην πρόταση των κοινών διατάξεων. Συνεπώς, στην απάντησή μας, στην πρόταση, αναφερόμαστε ακόμα περισσότερο στην αρχή έτσι ώστε να μπορέσουν να προκύψουν περισσότερα αποτελεσματικά ουσιαστικά δικαιώματα για τους Ευρωπαίους. Από αυτή την άποψη θα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο από να επιδιώξουμε τους στόχους αυτής της πολιτικής. Δηλαδή εργασίες και ανάπτυξη. Αν θέλουμε όμως να προσεγγίσουμε όλους τους Ευρωπαίους, χρειαζόμαστε κοινωνική και οικονομική σύγκληση. Η κοινωνική ένταξη θα πρέπει επίσης να είναι ένα στόχος και να έχω συμπεριλάβει στην πρόταση. Παρ' όλα αυτά, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τη σύγκληση μεταξύ της Ανατολής, της Δύσης, του Βορρά και του Νότου, κατά την άποψή μου είναι αναγκαίο να υπάρξει μία αύξηση της ε, του προπολογισμού συνοχής. Κατά την άποψή μου αυτό είναι ζωτική σημασία και κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρχει ένα μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού για το τομέα αυτό. Ε, για να είμαστε σίγουροι ότι τα ποσά αυτά θα μπουν κατά μέρος ε, σε επίπεδο κάθε χώρα. Αυτό μου ε, οδηγεί στο επόμενο σημείο. Όταν συγκρίνουμε την πρόταση της Επιτροπής με την τρέχουσα πρόταση, την, ε, την συγχρηματοδότηση και την προχρηματοδότηση, θα δούμε ότι αφορά ορισμένες περιοχές ε, για να μην παρεμποδίσουμε την εκτέλεση των προγραμμάτων σε επίπεδο κρατών μελών. Προτείνουμε την αύξηση του ποσοστού προχρηματοδότησης και συγχρηματοδότησης. Διαφορετικά θα υπάρχει ένα κατόφλι για αυτές τις περιφέρειες που περισσότερο χρειάζονται τα κονδύλια. Τώρα, κάτι περισσότερο για τη χρηματοδότηση από την Ευρώπη. Επιτροπή ε, ε, η για μεγαλύτερη συνοχή σε ό,τι αφορά τη χρήση των κοινοτικών ταμείων και των συγκεκριμένων συστάσεων των χωρών. Στην πρότασή τους τα κονδύλια θα πρέπει να καταβάλλονται μόνο σε περίπτωση που γίνονται οι απαραίτητες ε, μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να την υπόψη και οι προκλήσεις όπως έχουν εντοπιστεί στους κοινωνικούς πίνακες αποτελεσμάτων καθώς και στην κοινή ε, ε, έκθεση και θα πρέπει να ε, τροποποιούνται ανάλογα για να μπορέσουν να αντικατοπτρίσουν αυτή την ανάγκη. Σε περιπτώσεις που θεωρείται ότι θα πρέπει να ληφθεί διορθωτική δράση, θα πρέπει τη έκθεση να λαμβάνεται υπόψη, δηλαδή η έκθεση για τον κοινωνικό, με τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων και να ε, υπάρχει, να είμαστε σίγουροι ότι λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις καθώς και ο κοινωνικός πίνακας και η κοινή έκθεση απασχόλησης είναι απαραίτητο προκειμένου οι κοινωνικοί εταίροι να διαδραματίσουν ρόλο στην διαμόρφωσή του και ενώ οι χώρες μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν για το περιεχόμενο. Αντιδρώντας ε, λοιπόν στην πρόταση της Επιτροπής, πιστεύω ότι θα πρέπει να ενδυναμωθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Τελειώνοντας, ε, θα ήθελα να πω ότι ότι η καλύτερη προσβασιμότητα στα ταμεία είναι σημαντική για να υπάρξει καλύτερη απορρόφηση. Είμαι υπέρ της μείωσης του διοικητικού άγχους και της αύξησης της ευελιξίας. Θα πρέπει βεβαίως να κάνουμε ορισμένες ρυθμίσεις στην πρόταση για να προκύψει περισσότερη ελληνική και πραγματικά ανυπόμονα περιμένω να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους κοιόδες εισηγητές, ξεκινώντας από το ΕΛΚ και τον κύριο Σόγκορ. Σας ευχαριστώ. μια ενισχυμένη και με περισσότερη εστίαση πολιτική συνοχή θα επιτύχει σύγκληση σε όλε τι περιοχέ και σε όσο το δυνατόν περισσότερε ομάδε ανθρώπων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα συμπεριλαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότεροι ε, άνθρωποι στι ε, νέες έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στι νέε προκλήσει τη κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση τη Κομισιόν είναι πάρα πολύ καλή και καταφέρνει να συμφιλειώσει τι διάφορε ανάγκε, ξεκινώντα από του δημοσιονομικού περιορισμού ε, που θα επιφέρει το Brexit, ε, συμφιλιώνοντας την ανάγκη για λογοδοσία, τι νέε αναδυόμενε προκλήσει και τι απαιτήσει των διαφορών ενδιαφερόμενων φορέων. Στηρίζουμε λοιπόν την ε, κατεύθυνση που δίδεται τους στόχους της πολιτικής συνοχής στην προώθηση του πίνακα κοινωνικών επιδόσεων και του κοινωνικού προγραμματισμού, την επίτευξη ισορροπίας έτσι ώστε ε, να διατηρηθεί η οικειοποίηση στα κονδύλια και στηρίζουμε την πρόταση για αύξηση ορισμένων κονδυλίων στα πλαίσια του, του, του Επίσης, πιστεύουμε ότι χρειάζονται περισσότερες συζητήσεις μετά την ε, υποβολή των τροπολογιών, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί η κοινωνική συνοχή στους στόχους κοινωνικής συνοχής στο άρθρο 4. Είναι χρήσιμο να υπάρχει η επιλογή ελάχιστου ποσοστού χρηματοδότησης για τις επενδύσεις στην ε, ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, έτσι ώστε να αντιπαρέλθουμε τον ήδη μειωμένο προϋπολογισμό. Χρειάζεται επίσης να δούμε τις ανάγκες των επιμέρους κρατών μελών και το αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μπορεί να διατηρήσει μια ισορροπία. Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω και θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες έχει να κάνει με την πολιτική συνοχής και το Invest EU ε, το πρόγραμμα InvestEU δεν θα πρέπει να απορροφήσει κονδύλια που ε, χρειάζονται σε άλλους ε, νευραλγικούς τομείς. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στην ε, αγαστή συνεργασία με, τον, με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω τώρα εκ μέρου του κυρίου Γκέρικη από την ομάδα ECR, ο οποίο καλωσορίζει την πρόταση ε, ω απάντηση τη Ευρώπη στι ε, ανάγκε και απαιτήσει των πολιτών. Κατά τη διαβούλευση για τον κανονισμό όλοι οι φορείς συζήτησαν λιγότερους, σαφέστερους κανόνες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την υλοποίηση των ε, διαφόρων προγραμμάτων και τη χρήση των ευρωπαϊκών ε, ταμείων. Η χρήση αυξα... πρέπει να αυξηθεί και ταυτόχρονα η γραφειοκρατία να μειωθεί. Χρειάζεται να γίνονται σεβαστές οι ανάγκες των επιμέρους κρατών μελών και θεωρούμε ότι οι πέντε βασικοί στόχοι είναι αρκετά ισορροπημένοι. Ο εισηγητή τονίζει τη σημασία της ε, κοινωνικής Ευρώπης και του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Χρειάζεται επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία της Ευρώπης και στην ευφυή οικονομική μετάβαση, η οποία θα γίνει σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και σε ε, τοπικό πρώτα περιφερειακό πλαίσιο. Αυτά από τον κύριο και Τώρα θα δώσω το λόγο στη, στους φιλελεύθερους, ε, τον κύριο Καλβέ Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω αγγλικά και θα τελειώσω στα ισπανικά. Για να μην ε, μας πάρει και ο ύπνος. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, την εισηγήτρια την Άγνες για το σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με το CPR. Εμείς συμμεριζόμαστε τους ίδιους στόχους σε ό,τι αφορά τον στόχο της πολιτικής συνοχής της Ένωσης. Η πολιτική μου ομάδα υποστηρίζει μια ισχυρή πολιτική συνοχή που να καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη, όλες τις περιφέρειες της Ένωσης με έναν ε, προπολογισμό που θα αντιστοιχεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες της Ένωσης όπως ε, γνωρίζουμε, η έλλειψη συνοχής είναι και οικονομικό πρόβλημα, όχι μόνο κοινωνικό. Εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ το κοινωνικό πρόβλημα, αλλά είναι και οικονομικό. Διότι είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματική μια κοινωνία που δεν διέπεται από συνοχή. Η πρόταση για μια νέα, και ένα νέο κοινό κανονισμό, ε, κοινών διατάξεων ε, είναι πολύ σημαντική διότι εδώ περιλαμβάνονται οι βασικοί κανόνε τη πολιτική συνοχή τη Ένωση, ε, μεταξύ των οποίων και το ESF Plus για την επόμενη επταετία. Είναι ένα σύμβολο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, όπως λέει και η συγκήτρια. Υπάρχει ο κοινός στόχος, ε, θα πρέπει να υποστηρίξουμε μια πιο κοινωνική Ευρώπη που θα υποστηρίζει τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση όπου βρισκόμαστε στο τέλο ε, τη θητεία μα και όπου τα κοινωνικά ζητήματα έχουν όλο και μεγαλύτερη σημασία με βάση ε, εν ενόψη μάλλον των ευρωεκλογών. Εδώ μιλάμε για προχρηματοδότηση και για συγχρηματοδότηση και τις διάφορες ε, και διάφορα ποσοστά που προτείνει η συγκέντρια θα τα εξετάσουμε προσεκτικά. Είναι σημαντικό να παραμείνει το ίδιο επίπεδο επένδυσης ε, σε όλα τα ταμεία. Η συγκήτρια επίσης προτείνει να τροποποιήσουμε τους οικονομικούς φακές στις διάφορες, διάφορες, διάφορες κατηγορίες ε, περιφερειών. Εγώ μπορώ να την υποστηρίξω εφόσον βέβαια αυτό γίνει στα πλαίσια της συμφωνίας του Μαΐου στο, δημο, στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Δηλαδή, επίσης η πολιτική συνοχή και το ευρωπαϊκό εξάμεινο και η διαδικασία ευρωπαϊκού εξάμεινου θα πρέπει να συνδέονται όταν προγραμματίζουμε ε, τα ταμεία του ESI ε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αναμένω τη συνεργασία μας ε, για το σημαντικό, αυτό το σημαντικό κανονισμό και θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες για να βελτιωθεί περαιτέρω η πρόταση. Πάντως είναι πολύ καλή η βάση της πρότασης αυτής και τώρα θα περάσω στα ισπανικά διότι συνδέεται αυτό που θα πω με κάποιες χώρες ε, όπως η δικιά μου. Θα πρέπει να δούμε με την εισηγήτρια και τους συναδέλφους τι μπορούμε να κάνουμε εδώ, σε αυτό το κείμενο, για να βελτιώσουμε την ανάλυση εκ των υστέρων, την ex post ανάλυση των αποτελεσμάτων, την αποτελεσματικότητα, όχι ε, και βεβαίως και την ομιμότητα της χρήσης, ε, της ορθής ε, χρήσης των κονδυλίων βεβαίως. Αλλά ακόμα και εκεί όπου είχαμε ορθή χρήση, ποιο ήταν πραγματικά το αποτέλεσμα, ο αντίκτυπος σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Και να δούμε και αυτό το θέμα το οποίο βρίσκουμε ξανά και ξανά μπροστά μας. Κάποια χρήματα τα οποία τελικά δεν χρησιμοποιούνται. Σε συγκεκριμένες χώρες, σε συγκεκριμένες περιφέρειες συστηματικά. Κάτι δεν πάει καλά. Και θα πρέπει να το αναλύσουμε. Εγώ θα προσπαθήσω, αν μου το επιτρέπετε, διότι ο καθένας εδώ έχει τις δικές προθέσεις, να κάνουμε και μια αξιολόγηση ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα ε, σε οικονομικό κοινωνικό επίπεδο αν έπιασαν τόπο, προς τα χρήματα αυτά ε, και βεβαίως και η αρχική κατανομή ήταν σωστή. Αν, να δούμε λοιπόν αν ε, είχαμε πραγματική χρησιμοποίηση των κονδυλίων αυτών, διότι κάποιοι ε, χαίρονται όταν του χορηγεί τη χρηματοδότηση, αλλά όταν δεν φτάνει ποτέ στα χέρια του μετά δεν έχει νόημα. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Μπόιλαντ έχει το λόγο. Thank you, Chair. And first of all, Καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο γνωμοδότηση. Θα ήθελα να στήσω συγγνώμη επίση εκ μέρου τη κοιόδους εισηγήτριας Ειρήνα Κάρη που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, οπότε θα διαβάσω εγώ τα σχόλιά τη για την ε, Γκουε. Εμεί καλωσορίζουμε το γεγονό ότι επικεντρώνεται στην κοινωνική ένταξη η συγκήτρια, καθώ και την συμπερίληψη τη σύγκληση, τη αλληλεγγύη και τη συνοχή στο συνολικό στόχο αυτού του κανονισμού αργότερα στην Επιτροπή μας θα γίνει μια συζήτηση για την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές στην, στην ζώνη ευρώ. 120 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον γενικό αποκλεισμό. Έτσι λοιπόν η ομάδα μας συμφωνεί με την εισηγήτρια και την πρόθεσή της να αυξηθεί ο προπολογισμός για, για το Ταμείο Συνοχής και το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής Plus που παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης ε, βλέπουμε θετικά την προσπάθεια της ε, συγκίτρια να συνδέσει τα ταμεία με τον πίνακα αποτελεσμάτων τον κοινωνικό θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφέστερα, να αποτυπώνεται σαφέστερα οι αρχές του πυλώνα ε, κοινωνικών δικαιωμάτων. Δεν θέλουμε από εκεί πέρα να συνθούν περαιτέρω τα ταμεία αυτά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τις σχετικές συστάσεις αναχώρα που συνήθως αντιβαίνουν ε, τον στόχο της κοινωνικής συνοχής και τα συμφέροντα των εργαζομένων. Επίσης είμαστε κατά των μακροοικονομικών προϋποθέσεων που επιτρέπουν στην Κομισιόν να σταματήσει την πληρωμή όταν δεν υπάρχει ε, συμμόρφωση με την δημοσιονομική πειθαρχία. Επίσης δεν μπορούμε να, να υποστηρίξουμε την, ε, το, το Ταμείο InvestEU, ε, διότι ουσιαστικά μας οδηγεί στο να περάσουμε από ενισχύσεις σιγά σιγά σε δάνεια ε, αναμένουμε με ενδιαφέρον τις μελλοντικές συζητήσεις για αυτόν τον κανονισμό. Ευχαριστώ. Και τώρα για τους πράσινους η κυρία Βάνε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την κυρία εισηγήτρια για την παρουσίαση της γνωμοδότησής της. Θα ήθελα και να συμφωνήσω απόλυτα με όσα λέτε για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, διότι και εμείς είμαστε της άποψης ότι η πολιτική συνοχή γενικότερα και τα ε, διαρθρωτικά ταμεία ειδικότερα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο επίδειξης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για τις περιφέρειες, για ε, τα κράτη, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, της φτώχειας και πολλών άλλων. Στη, σε διάφορες εκθέσεις ε, που αφορούν τη συνοχή έχουμε δει ότι δημόσιες επενδύσεις ε, είχαν προβλήματα σε αρκετές περιφέρειες, ιδιαίτερα επενδύσεις ε, οι οποίες ήταν αναγκαίες. Χωρίς λοιπόν αυτά τα ταμεία και χωρίς την πολιτική συνοχή δεν θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί. Αυτό μας δείχνει πόσο σημαντικά είναι. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι πέραν από τόσα επικίες και με τα οποία συμφωνώ θα... Ε, έχουμε και εμείς τις δικές μας προτάσεις. Μία από αυτές αφορά το Invest EU στο άρθρο 10. Ε, δεν συμφωνούμε με αυτήν την πρόταση, διότι υπάρχει διαδικασία omnibus ε, κατά της ε, δυνατότητας μεταφοράς κονδυλίων και αυτό μας φαίνεται πως είναι μία επίθεση κατά της πολιτικής συνοχής. βλέπουμε ότι από το ΕΦΣΙ ελάχιστα κονδύλια πηγαίνουν προς την ε, πολιτική συνοχής. Γι' αυτό λοιπόν ε, όσα έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε μετά από πολύ αγώνα, όπως για παράδειγμα τα κονδύλια για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής του περιβάλλοντος, με την πρόταση αυτή θα εξαφανιστούν, θα τα χάσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ την προσέγγιση αυτή λάθος. Μετά, Αναφέρθηκε ήδη το ότι υπάρχουν ανησυχίες για τα χαμηλά ποσοστά συγχρηματοδότησης. Ε, δεν αφορούν μόνο ε, περιφέρειες αλλά και οργανισμούς οι οποίοι δεν ε, έχουν καθόλου πρόσβαση στα ταμεία, στη χρηματοδότηση. Άρθρο λοιπόν 106 Εδώ θα υποβάλουμε τις δικές μας τροπολογίες για τις μακροοικονομικές προϋποθέσεις και την μεγαλύτερη σύνδεση με την οικονομική δικυβέρνηση. Είμαστε κατά αυτών. Όχι μόνο επειδή το θεωρούμε βασικά δομικά λάθος ε, το ότι τιμωρούνται δηλαδή οι περιφέρειες όταν δεν επιτυγχάνουν ορισμένους στόχους αλλά επειδή ασκείται πίεση λόγω της πολιτικής ε, λιτότητας ε, στους ε, δημόσιους προϋπολογισμούς, κάτι το οποίο θεωρούμε θεμελιωδώς λάθος. Μετά, η επαναχρησιμοποίηση των οριζόντιων αρχών είναι κάτι που θεωρούμε πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα η απαγόρευση των διακρίσεων. Ε, αυτό βρίσκεται στις αιτιολογικές σκέψεις και θεωρούμε πως χρειάζεται να προβληθεί περισσότερο. Μετά, ε, θα πρέπει να αναφερθούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κυρία εισηγήτρια η ανέφερε πολύ σωστά ε, την ενίσχυση των κοινωνικών εταίρων σε όλη την διαδικασία. Ε, και εμείς επιθυμούμε μεγαλύτερη συμμετοχή των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων, για παράδειγμα, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει κάποιος από το EFTD, από το ENF, γι' αυτό λοιπόν θα δώσω το λόγο στην κυρία Μωράν Σαχτιέ και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτού λάβει ξανά το λόγο η συγγήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την ε, Άγνες Γιουγκέριους που έκανε μια πολύ καλή ε, γνωμοδότηση στο όνομα της Επιτροπής μας για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση που μας υπέβαλε. Εξαιρετικά σημαντική και αυτή βρισκόμαστε εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης. Βλέπουμε ότι όλα τα χρήματα, όλα τα κονδύλια που μπορούμε να κινητοποιήσουμε για να μπορέσουν οι άνθρωποι να παραμείνουν στον, στην αγορά εργασίας και να τους προετοιμάσουμε για τις εξελίξεις στον χώρο εργασίας είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο λοιπόν που θα πρέπει να μας κινητοποιεί είναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες που αυτή τη στιγμή εργάζονται θα πρέπει συνεχώς να είναι προσπαρμοσμένοι στι εξελίξεις της εργασίας τους. Πρέπει να είναι ένας πολύ σημαντικός άξονας της χρησιμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε, να προετοιμάσουμε τους ανθρώπους αυτούς δηλαδή ε, για τις εξελίξεις στον χώρο εργασίας τους. Είναι δηλαδή ένα ταμείο ε, που θα βοηθάει τους τρόπου αυτούς να προσαρμοστούν. Κάτι άλλο τώρα που είπαν και οι συνάδελφοι. Η απλοποίηση. Η διευκόλυνση της πρόσβασης. Η Επιτροπή έχει υποβάλει μια σειρά από προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Παντού, όταν μιλάμε με τους ανθρώπους, τους ενδιαφερόμενους, μας λένε είναι πολύ περίπλοκη διαδικασία. Πρέπει να μπορούμε να πλουστεύσουμε τα πράγματα. Αυτό σημαίνει όμως ε, ε, ότι θα πρέπει τα διάφορα έγγραφα που προτείνονται εμείς να τα πετσοκόψουμε διότι όλα τα project έχουν ενδιαφέρον και τα μικρά και τα μεγάλα. Θα πρέπει λοιπόν να απλουστεύσουμε την προσβασιμότητα και να προσθέσω ότι θα πρέπει να απλουστεύσουμε και τους ελέγχους. Κάτι που συχνά μας προσάπτουν είναι ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία φτάνουν όταν πια έχει ολοκληρωθεί το project. Για κάποιες μη κυβερνήσεις οργανώσεις, για κάποιες ε, ε οργανώσεις, ε, είναι δύσκολο να βρουν τα χρήματα στην αρχή. Πρέπει να έχουν ένα κεφάλαιο αρχικό. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει, Άγνες, αυτό να αποτυπώνεται στην έκθεση. Είναι σημαντικό. Διότι ουσιαστικά χάνουμε κάποια project. Συχνά έχουμε ένα καλό project, αλλά δεν υπάρχουν τα χρήματα για να το υποστηρίξουν αρχικά. Αυτό ήθελα να το υπογραμμίσω. Τέλος, το πρόβλημα του χρονοδιαγράμματος. Ακούω κάποιους εδώ ε, που κάνουν πολιτική και λένε Α, αυτά τα ταμεία θα τα δούμε μετά τις ευρωεκλογέ. Όχι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει ούτως ή άλλως καθυστέρηση στην αφετηρία. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι τους κανόνες του παιχνιδιού για να μπορέσουν ήδη από τώρα στην αρχή της περίοδου να προετοιμάσουν τα project τους. Και εγώ ε, περασπίζουμε με νύχια και με δόντια να σταθεροποιήσουμε τώρα τα κονδύλια από τα ταμεία αυτά, ιδάλλως θα αργήσουμε πολύ και θα πάμε στο 21, το 22, το 23. Δεν δείχνει έτσι η Ευρώπη την αποτελεσματική. Και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και σε όλα αυτά τα ταμεία συνοχής είναι η πραγματική αποτελεσματικότητα, ο πραγματικός αντίκτυπος επιτόπου. Πέρα νομίζω από τις όποιες ε, πολιτικές διαφορές μπορεί να έχουμε, νομίζω πως αυτά τα τέσσερα σημεία μας βρίσκουν σύμφωνους και θα πρέπει να τα προωθήσουμε. Και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ε, Άκνες, ε, η οποία γνωρίζω ότι θα επιμείνει μέχρι τέλους. Σας, σας ευχαριστώ κυρία Σουκβά, Γενική ε, Υποδιευθύντρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι μας βρίσκει σύμφωνος η έκθεση της κυρίας Κιονγερίωσα προκειμένου να υπάρξει αυτός ο κανονισμός η Επιτροπή πρότεινε μια κοινή αντίληψη για το Ταμείο Συνοχής για το 2020 Βεβαίως με μια απλοποίηση των κανόνων και των διαδικασιών. Συμφωνούμε με τους συνομοθέτες για έτσι ώστε να μπορέσουν να προκύψουν περισσότερα ωφέλη από τις πολιτικές συνοχής. Λαμβάνουμε υπόψη μας το γεγονός ότι θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν όλα αυτά με τα κοινωνικά δικαιώματα και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κάναμε μία επιλογή συγκεκριμένων κανόνων που μπορούν να εφαρμοστούν οριζόντια και στα επτά ταμεία, στον κοινό κανονισμό για την εφαρμογή των πέντε στόχων. Ο στόχος 4 για περισσότερο κοινωνική Ευρώπη είναι το φυσικό όχημα για την εφαρμογή όλων αυτών Οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί δείχνουν ε, την πρόθεσή μας για επίτευξη των στόχων με μία ενισχυμένο προπολογισμό. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα από τα βασικά σημεία συζήτησης στα, στο πολιτείας πλαίσιο και πιστεύουμε ότι ο προϋπολογισμός που προτάθηκε από την Επιτροπή παρουσιάζει με έναν ρεαλιστικό τρόπο το μέλλον του προπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη το Brexit και τις επιθυμίες των κρατών μελών. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη τα όσα υπόθηκαν για την προχρηματοδότηση και τη συγχρηματοδότηση. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι μία πρόθεση να κρατηθεί το επίπεδο επενδύσεων στο ίδιο επίπεδο σε ό,τι αφορά την προχρηματοδότηση. Αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα του προπολογισμού. Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία που θα αποτελέσουν θέμα συζήτησης μεταξύ των σύνομοθετών. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πολιτικής ενοχής η, πολιτική, η Επιτροπή προτείνει ένα πάγιο ποσό 100 εκατομμυρίων και πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι θετικό σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες και τις προτεραιότητες που θέτει η Επιτροπή για το μέλλον. Στόχος δηλαδή είναι η επένδυση των ε, στους ανθρώπους. Πιστεύουμε ότι η ευελιξία που προτείνεται στον κανονισμό για μια μεταφορά μεταξύ των ταμείων μέχρι 5% σε, χώρε, χώρες μέλη που θέλουν να, περάσουν αυτό το επίπεδο και να το αυξήσουμε ένα επιπρόσθετο 5% είναι μια δυνατότητα για όλους. Επίσης, καλωσορίζω την αναφορά στην υιοθέτηση του κανονισμού πριν από τις εκλογές. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ευκρίνεια και θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να διαπραγματευτούν με την Επιτροπή και να υιοθετούν τα προγράμματα έγκαιρα. Συνεχίζουμε να είμαστε φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά αυτό. Έχουμε απόλυτα ξεκάθαρες απόψεις και επιθυμούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι έγκαιρα προετοιμασμένα. Βεβαίως, περιμένουμε τις δικές σας απόψεις. Thank you. Uh, Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην εισηγήτρια. Μόνο δύο λόγια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλες ε, τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους συναδέλφους Βεβαίως είμαι αναμονή των προτάσεών τους. Πιστεύω ότι θα το πείτε κι εσείς ότι η προθεσμία είναι στο τέλος της εβδομάδας για την κατάθεση των τροπολογιών. Απαντώντας στα όσα είπατε εσείς, ε, εκπροσωπώντας την Επιτροπή, θα ήθελα να πω ότι και εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το να υπάρξει σαφήνεια σε ό,τι αφορά τους νέους κανόνες και τον κανονισμό σε όλα τα κράτη-μέλη και στα, στις ε, ΜΚΟ και αυτό να γίνει πριν από τις επόμενες εκλογές. Αυτά είναι προγράμματα τα οποία θα πρέπει να γίνονται στις διάφορες χώρες μέλη. Και πιστεύω ότι θα είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί αυτό το συντομότερο δυνατόν. Ακούω όμως ότι όλοι ενδιαφέρονται να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση και περιμένω λοιπόν τους επόμενους μήνες για να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 28 Σεπτεμβρίου 2018 στις 12 το μεσημέρι. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η συγγήτρια είναι εδώ. Πολύ ωραία. Θα δώσω λοιπόν το λόγο αμέσως στην κυρία Κλούν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, να πω πως ε, στηρίζω απόλυτα την πρωτοβουλία. Είναι μια εξαιρετική πρόταση για τους νέους Ευρωπαίους πολίτες και για τις κοινότητες επίσης, ε, με την οποία οι πολίτες μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε διάφορα προγράμματα αλληλεγγύη σε όλη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα γνωρίζουμε ότι ήταν επιτυχές, έχει ενώσει τους νέους, έχει φροντίσει προ τη δημιουργία μια κοινωνίας χωρίς αποκλεισμού και έχει αντιμετωπίσει μία πληθώρα από προκλήσεις. Η πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλοδεχούμενη. Βλέπουμε ότι η έμφαση δίνεται στην αλληλεγγύη και δίνονται δυνατότητες στους νέους να την εκφράσουν. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία δεξιοτήτων που θα μπορούν να μεταφερθούν μετά με τη σειρά τους στην αγορά εργασίας και ε, να ε, αυξήσουν ε, την απασχόληση και οι νέοι θα έχουν την δυνατότητα να πάνε σε διάφορες κοινότητες, να εργαστούν και να συνεισφέρουν με τρόπο που θα βοηθήσει τις ε, πόλεις αυτές, τις κοινότητες ή τις περιφέρειες, μαθαίνοντας ταυτόχρονα νέες δεξιότητες ή αναπτύσσοντας τις υπάρχουσες. Στο σχέδιο γνωμοδότησης θα ήθελα να επαναλάβω λοιπόν ότι ο εθελοντισμός και η μαθητεία δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την αμοιβόμενη εργασία και δεν πρέπει να θεωρείται ε, πως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και θα ζητήσουμε λοιπόν συμμετοχή των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων σε ε, πλατφόρμες όπου μπορούν να ε, διερευνήσουν το πώς μπορεί να γίνει η πρόσβαση των νέων στην πιο εύκολη. Σε ό,τι αφορά τις μαθητείες, θα πρέπει να υπάρχει ένα κομμάτι που θα διασφαλίζει υποστήριξη διοικητική, γλωσσική και ποιοτική και θα ζητήσουμε να δοθεί έμφαση στο πλαίσιο ποιότητας για τη μαθητεία. Θέλουμε να μπει στην κορυφή των προτεραιοτήτων και θα το ζητήσουμε αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι θεωρούμε ότι οποιαδήποτε μαθητεία που προσφέρεται θα πρέπει να ε, ενστερνίζεται αυτές τις ε, αξίες και τις αρχές. Την τελευταία φορά που συζητήσαμε συζητήσαμε και για τη χρηματοδότηση και θεωρούμε πως η χρηματοδότηση θα πρέπει να διανέμεται εξίσου και, στους, ε, τρεις, ε, και στις τρεις κατηγορίες του προγράμματος. Προσβλέπω λοιπόν στην ε, καλή συνεργασία με όλους τους σκιώδεις εισηγητές Γνωρίζετε ότι στην ε, Επιτροπή συζητήθηκαν ήδη πάρα πολλά που θα μας βοηθήσουν. Έχει συζητηθεί και το πρόγραμμα αλληλεγγύης. Γι' αυτό λοιπόν είμαι σίγουρη πως αυτές οι συζητήσεις θα συνεχίσουν και στο μέλλον και θα είναι επιτυχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Γιονκέριου εκ μέρου των ε, Σοσιαλδημοκρατών. Μάλιστα. Μου φαίνεται πω ο σκιώδη εισηγητή ε, είναι στι Βρυξέλλε, αλλά δεν έχει καταφέρει να βγει από το αεροπλάνο. Δεν ξέρω λοιπόν τι έχει συμβεί. Μου ζήτησε όμω να διαβάσω το μήνυμά του. Λέει λοιπόν ο συνάδελφος ότι θα ήθελε καταρχάς να ευχαριστήσει την ε, κυρία εισηγήτρια, την κυρία Κλούν για την ε, γνωμοδότηση ε, στην πρόταση. Πολλές από τις απόψεις του είναι και απόψεις αυτής της Επιτροπής οι οποίες έχουν διατυπωθεί ήδη μερικούς μήνες πριν όταν συζητήθηκε η νομική βάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο θα ε, τρέχει μέχρι και το τέλος ε, του φυστάμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαίσιου μέχρι το 2021. Ή, ίσως θυμάστε ότι ο κύριος Μπρόντο ως... Ε, σκιώδη εισηγητής, μαζί με τη συνεργασία τη, συζητήρια και των υπόλοιπων σκιωδών, κατάφερε να επιτύχει πολύ θετικά αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, οι οποίες ήταν ε, δυσκολίες κυρίως σε διαδικαστικά θέματα και στη συνεργασία με Συμβούλιο και Επιτροπή. Μου ζήτησε λοιπόν ο συνάδελφο να, να σας πω ότι εξαιτία όλων αυτών η κυρία Κλούνθα αναλάβει το θέμα αυτό, μια και γνωρίζει πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Το κάθε τεχνικό στοιχείο, την κάθε λεπτομέρεια, μια που συμμετείχε στην ανταλλαγή απόψεων και είναι σίγουρος πως η συνεργασία θα είναι εξαιρετική όπως ε, άλλωστε ήταν και στο παρελθόν. Και είναι σίγουρος επίσης ότι θα βελτιωθεί το κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από τις ε, συζητήσεις στην Επιτροπή. Ο συνάδελφος θεωρεί ότι το κύριο μήνυμα της γνωμοδότησης της Επιτροπής μας θα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πρέπει να είναι ένα μέσο που θα δημιουργεί ποιοτικέ προτάσεις και απτά πραγματικά ωφέλη σε πολλούς ε, που χρειάζονται βοήθεια στην Ευρώπη και πώς ε, θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους να ε, συνεισφέρουν θετικά προς όφελος των συμπολιτών τους. Είναι σίγουρος πως ε, το πρόγραμμα είναι φιλόδοξο και θα είναι αρκετά ποιοτικό και θα ήθελε λοιπόν να εκφράσει τη στήριξή του σε οποιαδήποτε πρόταση ακολουθεί την κατεύθυνση αυτή, της βελτίωσης δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν και οι κατευθυντήριες γραμμές ε, είναι προτάσεις τις οποίες μπορεί να στηρίξει και ελπίζει να στηρίξει και η Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και σας εύχεται καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι σκιώδη συγκήτρια για την ομάδα ECR και θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να φορέσετε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Μπορώ να συμφωνήσω με πολλά ε, σημεία της γνωμοδότησης και στις δικές μου τροπολογίες θα δώσω έμφαση σε δύο τομείς που θεωρώ πολύ σημαντικούς. Πρώτα, θεωρώ πως θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στο εξή. Όλες οι δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και ενώ όλες θα είναι προσβάσιμες σε όλους, δηλαδή και στα άτομα με αναπηρία και σε άτομα ε, με διάφορες άλλες ε, δυσκολίες. Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν, ιδιαίτερα σε άτομα με αναπηρία, να συμμετέχουν συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία για το δωρεάν εισιτήριο ε, Interrail στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν οι νέοι αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα μετά τα 18 τους χρόνια να αποκτήσουν ένα τέτοιο εισιτήριο για να ταξιδέψουν. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να κάνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ξεχνά τα άτομα με αναπηρία, ιδιαίτερα τους νέους με αναπηρία. Διότι έχουν ειδικέ ανάγκες ε, στα ταξίδια για παράδειγμα. Χρειάζονται υποστήριξη ιδιαίτερε εγκαταστάσει, ε, προσαρμοσμένες εγκαταστάσει. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τα άτομα με αναπηρία και να τους παρέχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν και εκείνοι σε όλα αυτά τα project. Χρειάζεται λοιπόν να φροντίσετε τη συμπερίληψη και αυτής της ομάδας ανθρώπων. Τώρα ε, θα... Ε, ήθελα να σας ενημερώσω επίσης ότι θα επικοινωνήσω με τον Επίτροπο Ναύρατζιτς μάλλον επικοινώνησα με τον Επίτροπο και τον ρώτησα πόσοι από αυτούς τους ε, νέους χρησιμοποίησαν αυτή τη δυνατότητα του δωρεάν εισιτηρίου και μου είπε ότι από τις 15.000 ε, μόνο 7.500 μόνο 27.000 μάλλον Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσει αυτή η πρωτοβουλία διότι οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια να ενημερώνονται καλύτερα οι νέοι ιδιαίτερα οι νέοι που έχουν διάφορα προβλήματα υγείας ώστε να μπορέσουν να ε, συμμετέχουν σε αυτά τα project. Αυτό ήταν ένα μόνο παράδειγμα έτσι ώστε να καταστεί σαφές ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει και εκείνα να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής. Χρειάζεται λοιπόν να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή. Γι' αυτό και θεωρώ ότι στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και έμφαση στα άτομα με αναπηρία από ό,τι προηγουμένως. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω χρειάζεται να δοθεί προσοχή στην ε, επιστοποίηση των διάφορων δεξιοτήτων, ε, δυνατοτήτων, οι οποίες πρέπει να ε, αναγνωρίζονται εγγράφως. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω και εγώ σε μια καλή συνεργασία. Θα περάσουμε τώρα στην ομάδα των φιλελεύθερων. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποιος. Η κυρία Μπόιλαν παρακαλώ για την Γκούε. Ναι, ευχαριστώ και πάλι. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια, την κυρία Κλούν, για την γνωμοδότηση. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ε, έχει κάποια προβληματικά στοιχεία. Η συμπερίληψη ε, των, ε, των, του τομέα του κερδοσκοπικού ε, μπορεί να οδηγήσει στο να εργάζεται κόσμος δωρεάν ε, για κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ε, το τελευταίο που χρειάζονται οι νέοι σήμερα είναι ένα πρόγραμμα που θα επιτρέψει ε, τους ε, κερδοσκόπους να τους εκμεταλλευτούν. Χαίρομαι που γίνεται μια αναφορά στο σχέδιο γνωματότηση ότι τα στάζ αυτά δεν εγκαταστούν ε, τις θέσεις απασχόλησης και ο ορισμός της απασχόλησης ως αμοιβόμενη δραστηριότητα ε, θα πρέπει να είναι σαφής. Να γίνει σαφής διαχωρισμός λοιπόν μεταξύ του εθελοντισμού και της ε, ε απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ουσιαστικά είναι σαν να παίρνουμε τα χρήματα από τη μία τσέπη και να τα βάζουμε στην άλλη. Παίρνουμε χρήματα από από προγράμματα που υπάρχουν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να χρηματοδοτήσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Θα πρέπει λοιπόν να, να βελτιώσουμε το υπάρχον πρόγραμμα εθελοντισμού και να μην δημιουργούμε ένα νέο πρόγραμμα και να υπονομεύουμε αυτά που υπάρχουν ήδη. Έτσι λοιπόν ε, είναι σημαντικό αυτός ο κανονισμός να περιλαμβάνει ένα σαφή κανονισμό του εθελοντισμού. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτικέ δυνατότητε εθελοντισμού που θα, που ε, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια αμοιβόμενη εργασία. Θα συνεργαστούμε με τους συναδέλφους ε, για να εξασφαλίσουμε ότι όντως αυτό θα αποτυπώνεται στο κείμενο. Ευχαριστώ. Και τώρα για τους πράσινους η κυρία Λάμπερτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, δεν ήμουν εδώ στην αρχή. Ε, ήθελα απλώς να πω ότι για μας αυτά που ελέγχθησαν για την ε, ε, διαφορετικότητα είναι πολύ σημαντικά. Εάν έχουμε αυτό το νέο ξεχωριστό πρόγραμμα, είναι σημαντικό να είναι διαθέσιμο ε, σε μια ευρύτερη γκάμα ανθρώπων, σε όσο γίνεται ευρύτερη γκάμα. Πρέπει η διάσταση της κοινωνικής ένταξης να ληφθεί υπόψη. Συμφωνούμε και με αυτό που μόλις ελέγχθη και αυτά που συμφωνήθηκαν στο κείμενο, ότι δεν πρόκειται εδώ για υποκατάστατο ε, μιας ε, αμοιβόμενης εργασίας, αλλά ως μια προετοιμασία για την απασχόληση. Και βέβαια υπάρχει το θέμα του προπολογισμού. Εδώ νομίζω το καταλάβαμε όλοι στην Επιτροπή αυτή. Παίρνουμε χρήματα από αλλού και μάλιστα από τομείς που χρειάζονται χρήματα και δεν δημιουργούμε μια ξεχωριστή νέα δημοσιονομική γραμμή. Βεβαίω είναι ε, χαμένη μάχη αυτή, αλλά θα πρέπει εμεί να πούμε ότι εδώ έχουμε νέα πρόγραμμα που χρειαζόμαστε και νέα χρήματα. Δεν μπορούμε να τα παίρνουμε από αλλού και να σαλαιμοποιούμε τι πολιτικέ μα και τα κονδύλια μα. Αναμένουμε με ανεπιμονησία τη συνεργασία με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ από την EFDD, την ENF δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος η κυρία Σόιντροβα τώρα έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Είμαι η συγκήτρια της Ευρωπαϊκής και Κοινωνική Επιτροπή, τη Κοινωνική Έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση για αυτόν τον νέο κανονισμό. Δεν γνωρίζουμε ή δεν έχουμε εν περιπτώσει κάποια ενημέρωση για την εφαρμογή. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν για μας να έχουμε κάτι τέτοιο, όμως ε, όλα αυτά θέλω να σε ευχαριστήσω για το σχέδιο γνωμοδότησης της συναδέλφου την κυρία Κλούν. Είναι πολύ καλό το κείμενο. Εκτιμώ ιδιαίτερα την προσέγγιση ε, για, τις, ε, το θέμα των δεξιοτήτων, ότι πρέπει η απασχόληση αλλά και ο να γίνει σε τομείς υψηλής ποιότητας ε, και να είναι προς όφελος των, τοπικών κοινωνιών και όχι υπέρ των ατόμων μόνο. Ε, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Εκτιμήσαμε επίσης το γεγονός ότι η κυρία Κλούν έχει ε, ενσωματώσει εδώ την ιδέα των πρέσβεων είναι σημαντικό για να αυξηθεί η ορατότητα αλλά και η προσβασιμότητα όπως ε, είπε και στην άλλη κυρία Τζιτνιάτσκα. Εάν θέλουμε ε, να φανούμε αντάξει της φιλοδοξίας ε, των ε, εκατοντάδων αυτών χιλιάδων θέσεων που θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, προτείνω οι εθνικοί οργανισμοί να ε, ενθαρρύνουν τους ε, συμμετέχοντες να είναι πρέσβεις για, αυτά τα προγράμματα. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να προχωρήσει αυτό. Αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή απασχόληση το θέμα της ε, επαγγελματικότητας και εγώ το σέβομαι αυτό. Από την άλλη είμαι πεπισμένη ότι ο εθελοντισμός πρέπει να είναι στην καρδιά και να είναι το βασικό κομμάτι της δραστηριότητας του συγκεκριμένου σώματος. Ε, ε, πρέπει να γίνει και μια κατανομή του προπολογισμού. Όμως, η κατανομή αυτή θα πρέπει να είναι ενδεικτική, έτσι ώστε να υπάρχει ευελιξία για να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί. Αυτό προτείνω. Τώρα, στην Επιτροπή Κούλτ έχω ήδη υποβάλει το σχέδιο γνωμοδότησης να αυξηθεί η, η ορατότητα του προγράμματος, να υπάρξει μια διαφοροποίηση στο σώστο προπολογισμό. Επίσης πρότεινα μια σειρά από τροπολογίες έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πνεύμα θελοντισμού στους νέους ανθρώπους μέσω του σώματος αλληλεγγύης, ε, να τους ενθαρρύνουμε να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες εθελοντισμού σε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Θα ήθελα επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων να εξαστούν τα ζητήματα ένταξης, διαφοροποίησης ανάλογα και με τη δραστηριότητα και να υπάρξει και ένας ορισμός της αλληλεγγύης να επανισάγουμε έναν ορισμό ε, για την αλληλεγγύη διότι στις διαπραγματεύσεις στον Τρίλογο υπήρχε ένας τέτοιος ορισμός θα υποβάλουμε ένα σχέδιο έκθεσης στις 10 Οκτωβρίου στην Επιτροπή μας και αναμένω να έχουμε μια καλή συνεργασία με τους συναδέλφους της Επιτροπής Απασχόλησης μιας και έχουμε τους ίδιους στόχους για να βελτιωθεί η κατάσταση των νέων. Ευχαριστώ και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Φραντς. Καλό σας απόγευμα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που μόλις είπε η κυρία Σόιντροβα σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση που υπάρχει. Οι διαπραγματεύσεις μόλις τελείωνα πριν από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη, υπάρχει στην ιστοσελίδα αλλά δεν έχει γίνει τίποτα σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις και τα προγράμματα. Ενδεχομένως αυτό θα γίνει αργότερα, στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Συνεπώς η πρόταση για το επόμενο πρόγραμμα σέβεται τις συμφωνίες που έχουν συναυτεί στις διαπραγματεύσεις με μερικές μικρές διαφορές συμφωνίες δηλαδή που έγιναν στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων γιατί η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση πριν την επίτευξη του τελικού της τελικής συμφωνίας. Θα ήθελα να πω και αυτό είναι μέρος των σχολείων που έχουν γίνει και στην Επιτροπή ΕΜΠΛ ότι υπάρχει κάποια διαφορά που βασίζεται στα όσα είπαν οι νομικέ υπηρεσίε. Έχουμε τα αναφέρει μερικές από τις παραγράφους που ήταν μέρος των ορισμών στο μέρος που αφορά τις δράσεις από τη στιγμή που δεν είναι ορισμοί αυτοί καθ' αυτοί, αλλά εξηγούν τους τρόπους των δράσεων που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Για παράδειγμα, το θέμα της εκμάθησης για την πρακτική και την εργαστία μπορεί ε, να το βρει κανείς στο άρθρο 8 του προτινόμενου κανονισμού. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν προτείνουν τον προϋπολογισμό και θέτουν τους στόχους για 350.000 νέους ανθρώπους που θα στηριχτούν από αυτό το 1,26 δις ε, ευρώ θα ήθελα να πω ότι σεβαστήκαμε τις συμφωνίες που έγιναν στις διαπραγματεύσεις στο κεφάλαιο που αφορά την ε, συμμετοχή των νέων ανθρώπων. Υπάρχουν κοινωνικές προκλήσεις. Στο κεφάλαιο 3, πόσο του κανονισμού, έγινε σεβαστό το 90% για τους εθελοντές και το 10% για άσκηση, για πρακτική άσκηση. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η πρόταση αυτή δεν είχε στόχο μόνο το να δημιουργήσει ε, το, ένα one-stop shop για τους νέους ανθρώπους σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη την διέπουν και δύο αρχές που τονίσαμε πάντοτε, η ποιότητα, η υψηλή ποιότητα των δραστηριοτήτων και δεύτερον την ένταξη. Εμείς βασιζόμαστε σε ένα άλλο παράδειγμα που δεν ανέφερε η προηγούμενη ομιλήτρια αυτό αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντών που έχει το 30% από τους ε, συμμετέχοντες. Δεν, εδώ δεν μιλάμε μόνο για νέους ανάπηρους, μιλάμε για νέους που δεν μπορούν ε, συνήθως να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες λόγω, για λόγους ε, ε, απόστασης από το κέντρο, για λόγους κοινωνικούς κτλ. Υπάρχει λοιπόν εντάχθηκε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και επιθυμούμε να εντάξουμε κάτι πέρα από τη χρηματοδότηση. Ελπίζουμε λοιπόν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη εμπλοκή των νέων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, ειδικά τα άτομα με ειδικέ ανάγκε και μπορούμε να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη είναι ένα πρόγραμμα για όλου. Ευχαριστώ πολύ. Η συγητή, η συγγήτρια τα ήθελα από δύο λόγια. Ωραία, δύο λόγια κύριε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσου πήραν το λόγο. Πραγματικά υπάρχει ένα κοινό πεδίο για όλου για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Είπατε κι εσεί ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι αυτή την εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντική και η παρέμβαση της ε, Επιτροπής Πολιτισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Επιτροπή και έχω την βεβαιότητα ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Okay, uh, Ένα σχόλιο να κάνω, επιτρέψτε μου. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 10 Οκτωβρίου. Ελπίζω να είστε σύμφωνοι με αυτό. Θα περιμένουμε τώρα λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε με το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ. Δεν So, dear colleagues, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να συνεχίσουμε. Η συγχύτρια για το επόμενο θέμα είναι εδώ, οπότε καθίστε σας παρακαλώ. Έτσι ώστε να συνεχίσουμε με τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διαιρέσεις. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην συγχύτρια. Κυρία Ανθία Μακιντάιρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά διότι η φωνή μου σήμερα είναι βραχνή, έχω βήχα, θα κάνω ό,τι μπορώ για να παρουσιάσω την έκθεσή μου. Έχει ζητηθεί λοιπόν να καταρτήσουμε γνωμοδότηση στην έκθεση αυτή Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι προς το παρόν η νομοθεσία έχει τεράστιες διαφορές από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και αυτό οδηγεί σε νομική αβεβαιότητα και αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν διασυνοριακά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό να καταπολεμηθεί και γι' αυτό χρειάζεται να επέλθει μία ε, συνοχή στην νομοθεσία στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ε, διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Θεωρώ επίση ότι οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι απλοί, ενιαίοι, σαφείς και ε, να μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα, να προστατεύουν ταυτόχρονα τον πολίτη αλλά και τις επιχειρήσεις και τους αλλά και τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών. Εφόσον οι κανόνες είναι ασαφείς ή δύσκολο να εφαρμοστούν, τότε πολύ πιθανό τα κράτη-μέλη να ερμηνεύουν διαφορετικά τους κανόνες αυτούς και ε, ως αποτέλεσμα μειώνεται η αποτελεσματικότητά τους και υπάρχει κίνδυνος κατακαιρματισμού της αγοράς. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να θεσπιστεί επαρκής προστασία για ε, τους ε, διάφορους ε, παράγοντας μιας επιχείρησης και τους υπαλλήλους ε, και να ε, θεσπιστούν μέτρα καταπολέμησης των, εταιριών, ε, των φαινομενικών εταιριών που είναι μόνο μια ταχυδρομική θηρίδα. Χρειάζεται επίσης τα μέτρα αυτά να είναι αναλογικά και όχι αποτρεπτικά για τους ειλικρινείς επιχειρηματίες που απλά θέλουν να επεκταθούν πέραν των συνόρων της χώρας τους. Χρειάζεται λοιπόν βελτίωση της ροής των πληροφοριών, της ε, συμβουλευτικής και της εκπροσώπησης ε, των εργαζομένων, αλλά χρειάζεται επίσης να φροντίσουμε οι απαιτήσει ε, να συνάδουν με την υφιστάμενη νομοθεσία. Καθώς ε, λοιπόν βρισκόμουν ε, σε στάδιο κατάρτισης της γνωμοδότησης προσπάθησα να ακολουθήσω όλα αυτά και να παραμείνω στους αρχικούς στόχους της οδηγίας ε, χωρίς να ξεφύγω από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Υπάρχει, από όσο γνωρίζω, μεγάλη στήριξη έτσι ώστε αυτή η οδηγία να διευρυνθεί και να καλύπτει και ε, την εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Συμφωνώ εν μέρη με αυτό, δεν ε, συμφωνώ όμως με το ότι αυτή η οδηγία είναι το κατάλληλο πλαίσιο για να ε, το χρησιμοποιήσουμε. Χρειάζεται φυσικά να γίνει εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης μια ευρύτερη συζήτηση, ε, δεδομένου ότι οι αναδιαρθρώσεις μιας εταιρείας έχουν επιπτώσεις στο ανθρώπινο εργατικό δυναμικό. Χρειάζεται γι' αυτό να γίνει μια πρώτερη ανάλυση. Ωστόσο, είμαι ανοιχτή για να συζητήσω με τους υπόλοιπους σκιώδεις το θέμα αυτό και να χρησιμοποιήσουμε προτάσεις σε περίπτωση μετατροπών όπου τα κράτη-μέλη θα χρειαστεί να διεξάγουν ενδελεχείς αναλύσεις σε μια εταιρεία εάν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι μια επιχείρηση εσκεμένα προσπαθεί να αποφύγει τις συνέπειες του νόμου ή να παραβιάσει νομοθεσία. Αυτό ισχύει στην περίπτωση των εταιρεών που είναι απλά νοματερίε που είναι με ταχυδρομική θηρίδα. Χρειάζεται λοιπόν να έχουν τη δυνατότητα οι αρμόδιες αρχές ε, να ε, παρεμβαίνουν και να διεξάγουν αναλύσεις για να διαπιστωθεί αν μια εταιρεία είναι τέτοια. Στην, ε, στις εκθέσεις που θα Γίνονται λοιπόν για αυτές τις ύποπτες εταιρείες βιτρίνες, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα αυτά υπόψη. Ο εισηγητής προσπάθησε να εναρμονίσει την έκθεσή του με την υφιστάμενη νομοθεσία, να συμπεριλάβει και το θέμα της διαβούλευσης με τους εργαζόμενους. Η οδηγια 2014, η οδηγία 2001 για τις μεταφορές και τις επιχειρήσεις και η οδηγία για τα συμβούλια εργαζομένων. Θα Χαρώ λοιπόν πολύ για την ανταλλαγή απόψεων που θα ακολουθήσει με τους και οδείς ε, Θα υποβάλουμε ορισμένες πρόσθετες τροπολογίες και θα χαρώ πολύ να συνεργαστώ με όλους τους σκιώδεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις, ξεκινώντας με τον κύριο Τσάμπα Σόγκορ εκ μέρους του ΕΛΚ. Okay. Thanks. Now working. Ναι, ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική η ελευθερία εγκατάσταση. Ε, Αναφέρει στην ενιαία αγορά, αλλά δεν υπάρχει, δεν έχει εφαρμοστεί πλήρω. Η άσκηση αυτή τη ελευθερία για τι εταιρείε παραμένει δύσκολη. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη τη ε, εισηγήτρια του για να μπορέσουν να εργαστούν αυτέ οι εταιρείε στην, στην ενιαία αγορά. Χρειαζόμαστε σαφεί, ενιαίου και εύκολα εφαρμόσιμου κανόνε. Επίση, πιστεύω ότι η πρόταση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε στο να διευκολύνει την διασυνοριακή κινητικότητα ε, βεβαίως σεβόμενοι τα ε, δικαιώματα των εργαζομένων, των ε, μετόχων, των επιχειρηματιών με τον ίδιο τρόπο και ισότιμα. Βεβαίω, όλα τα κρατημέλη δεν έχουν αυτό το σύστημα και τα μεταξύ των κρατών που το έχουν, οι κανόνε και πάλι ποικίλουν. Επιπλέον, οι κανόνε τη συμμετοχή των εργαζομένων με βάση την οδηγία για τι συγχωνεύσει ήταν απλησματική όπως λέει και η εξολόγηση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να επιβαρύνουμε περαιτέρω τι εταιρείε εφόσον δεν έχει αποδειχθεί ανάγκη για πιο περιοριστικέ απαιτήσει. Πέρα από αυτό θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο μεγαλύτερης απλούστευσης για να αποφύγουμε τις επικαλύψεις ε, σε ό,τι αφορά τις αναφορές και τις εκθέσεις. Αναμένω να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την εισηγήτρια και τους συνεισηγητές. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο κύριος Ντετιέν από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σα ευχαριστώ. πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμότατα την ε, κυρία Μακιντάρ για την γνωμοδότησή τη Αναμένω λοιπόν και εγώ την ε, συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων, διότι νομίζω πως η έκθεση αυτή αποτελεί μια εξαιρετική αφορμή γι' αυτό. Η έκθεση λοιπόν αυτή αφορά τις μετατροπές συγχωνεύσεις και διαιρέσεις, ωστόσο μένει αρκετός ε, χώρος για δημιουργική ε, νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Η ενίσχυση της κινητικότητας των επιχειρήσεων δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των εργαζομένων. Βλέπω πως ε, χρειάζεται επίσης ιδιαίτερα ιδιαίτερη προσοχή στις ε, διάφορες ε, διατάξεις Στην Γερμανία υπάρχουν πάνω από 50 εταιρείε με πάνω από 150.000 εργαζομένους. Γι' αυτό λοιπόν αυτό θέλει ε, προσοχή τα, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται και τα Συμβούλια Εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ε, δυστυχώς ε, υπάρχει μεγάλο, μεγάλος φόβος ε, για την απώλεια της ε, θέσης εργασίας κάποιου εάν συμμετέχει σε αυτά. Το άρθρο 86. Στην αρχική οδηγία είναι ένα άρθρο στο οποίο πιστεύω πως χρειάζεται πηγόντως βελτίωση. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, έχει παρουσιάσει καθώς φαίνεται ένα ισορροπημένο κείμενο, ε, έχει σοβαρές ελλείψεις σε ορισμένους τομείς. Δυνατότητα παγώματος ε, της δυνατότητας συναπόφασης συνεχίζεται, ε, δεν αλλάζει με την παρούσα πρόταση. Αυτό θα θέλαμε να αλλάξει, να αποτρέψουμε αυτήν ε, την ε, διάταξη προς όφελος των εργαζομένων. Χρειαζόμαστε ρυθμίσεις οι οποίες θα δίνουν ε, προστασία πάνω από το όριο των τριών ετών. Έχει συζητηθεί ήδη και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η συνάδελφος Ρέγνερ ζήτησε δέκαετη προστασία και συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Και επίσης ε, θα πρέπει να συζητήσουμε για τα ανώτατα όρια του αριθμού των ε, εργαζομένων πάνω από το οποίο θα, από το οποίο θα εφαρμόζεται η οδηγία. Θεωρώ πως η δική μας Επιτροπή πρέπει να εργάζεται προς όφελος των εργαζομένων και να φροντίσει για την προστασία αυτών. Επομένως, θα πρέπει να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε εντό των αρμοδιοτήτων μας έτσι ώστε να καταρτήσουμε μια γνωμοδότηση όσο το δυνατόν ε, ισχυρότερη που θα προσπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όμως και μακροπρόθεσμα ε, οφείλουμε να ε, κάνουμε πολλά για βελτίωση, να χρειάζεται να ενίσχυ, ενίσχυση της αυτονομίας των επιχειρήσεων και προστασία από οποιαδήποτε προσπάθεια καταστρατήγησης του δικαιώματος συναπόφασης των εργαζομένων στη Συμβούλια των Επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλντε Γκούε. υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος από αυτές τις πολιτικές ομάδες. Η κυρία Τζονγκερίους θα επιθυμούσε να πάρει το λόγο ή όχι. Μήπως η Επιτροπή θα ήθελε να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα. Επιτρέψα μου να πω δύο λόγια. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας, και αυτό είναι κάτι που έθιξαν όλοι οι ομιλητές, στη σημερινή συνεδρίαση, αυτό στο οποίο στοχεύαμε όταν υποβάλαμε αυτή την πρόταση, ήταν από τη μία πλευρά να δώσουμε στις εταιρείες τα μέσα για να μπορέσουν να αναδιαρθρωθούν διακρατικά και από την άλλη πλευρά να προστατεύσουμε αυτούς που χρειαζόντουσαν προστασία. Είναι σαφές ότι αυτός είναι ένας στόχος αυτής της Επιτροπής. διεξήχθησαν πολλές διαβουλεύσεις, αξιολογήθηκαν οι συνέπειες και πιστεύω ότι καταλήξαμε σε μια εξισορροπημένη πρόταση που καταφέρνει να συγκεράσει αυτούς τους δύο στόχους. Θα ήθελα να περιοριστώ στην απλή αναφορά των όπων όσο συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση αυτή που πιστεύω ότι είναι το βασικό μέλημα αυτής της Επιτροπής. Αυτό που προτείναμε δεν σημαίνει επανεφεύρεση του τροχού. Υπάρχει αναφορά στο υπάρχουν και εκτιμένο στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και στις ε, διακρατικές ε, συγχωνεύσεις. Υπάρχουν βεβαίως ορισμένα ε, σημεία προβληματικά. Αυτά τα σημεία αναφέρθηκαν από την ε, εκπρόσωπο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα ξεπερνώντας τα όσα ήδη υπάρχουν στο κεκτημένο. Για παράδειγμα, θέλουμε να κατόφλι για την συμμετοχή των εργοδοτών. Αυτό συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση που κάναμε. Επίσης, θελήσαμε να ενισχύσουμε το στοιχείο των διαπραγματεύσεων που υπάρχει στο κεκτημένο και σε ό,τι αφορά την τριετία Αναφερθήκαμε στην εταιρεία, ε, την τριετία κατά την οποία οι εταιρείε ε, δεν μπορούν να λάβουν μέτρα προκειμένου να υπάρξει συμμετοχή των εργαζομένων. Εκεί κάναμε μία αναφορά στα κεκτημένα περί συγχωνεύσεων. Θα ήθελα βεβαίως να πω, δεν σημαίνει ότι μετά από τρία χρόνια δεν θα υπάρχουν δικαιώματα και συμμετοχή των εργαζομένων, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι που σημαίνει ότι αυτή η περίοδος της τριετίας θα μπλοκάρει οποιασδήποτε μετέπειτα δράσεις της εταιρείας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι το υπάρχον και εκτιμένο για τις διαβουλεύσεις για την ενημέρωση των εργοδοτών είναι μη ε, ισχύων, δεν είναι είναι ανενεργό. Πιστεύουμε ότι προωθήσαμε ένα πακέτο το οποίο θα στείλει μήνυμα για συμμετοχή των εργαζομένων ιδιαίτερα ε, εκεί που έδειξαν οι διαβουλεύσεις ότι πρόκειται και ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα. Δεν θέλω να τελειώσω ευχαριστώντας την Επιτροπή που ανέλαβε αυτό το θέμα με τόση δεξιότητα Πιστεύουμε ότι θα ήταν σκόπιμο να επιτελεστεί πρόοδος έτσι ώστε να μπορέσουν πραγματικά να γίνουν ενεργοί όλοι οι κανονισμοί. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προηγούμενους ομιλητές για την θετική τους προσέγγιση. Περιμένω τη συνεργασία μαζί σας. Συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να δημιουργούμε κανόνες εκεί που χρειάζονται. Η απλοποίηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό συμφωνώ με αυτό που είπατε για τα τρία χρόνια και αυτό το θέμα ενδιέφερε ιδιαίτερα και την Επιτροπή. Αυτό που θα πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι αυτή είναι μια οδηγία που θα έχει ελάχιστα πρότυπα. Όλες οι χώρες μέλη μπορούν να προσθέσουν κάτι εδώ Ενδεχομένω σε ορισμένες χώρες θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω διευκρινήσεις. Ενδεχομένως δεν θα μπορέσουν όλα αυτά να εφαρμοστούν σε επίπεδο μικροδιαχείρισης. Αυτή είναι μία οδηγία και θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και να στοχεύσουμε σε κάτι το οποίο θα είναι αποτελεσματικό στη χρήση του. Ευχαριστώ. Σε 10 λεπτά, 10 λεπτά διάλειμμα. Ευχαριστώ.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

Καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Θα έλεγα να προχωρήσουμε με τα θέματα που μας απομένουν και στη συνέχεια να περάσουμε στην ψηφοφορία. Η έκθεση την οποία θα συζητήσουμε τώρα είναι η απασχόληση και οι κοινωνικέ πολιτικέ τη Ευρωζώνη. Ο κύριο Χέτμα είναι ο εισηγητή, δεν είναι εδώ όμω μαζί μα σήμερα. Η κυρία Κοσλόφσκα λοιπόν θα τον αντικαταστήσει. και υπάρχουν και τροπολογίε που έχουν υποβληθεί σχετικέ. κυρία Κοτλόσκα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να στείλω συγγνώμη στο όνομά του συναδέλφου που δεν μπόρεσε να είναι παρόν εδώ. Δεν μπόρεσε να φτάσει έγκαιρα και μου ζήτησε να διαβάσω την παρέμβασή του στα πολωνικά όμως. Οπότε βάλτε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ. Θα θυμάστε ότι η Επιτροπή μας ε, φέτος για πρώτη φορά είναι η αρμόδια Επιτροπή μαζί με την ΕΚΟΝ και αυτή τη στιγμή έχουμε κληθεί να εξετάσουμε το ρόλο της οικονομικής συμμετοχή των εργαζομένων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και επανένταξη των ανέργων. Είναι πολύ σημαντικά θέματα, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής πολιτικής διότι αφορούν ακριβώς την ανάπτυξη ε, της οικονομίας και την απασχόληση. Έχουμε εκατοντάδες ε, τροπολογίες, πολλές από αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, διότι κατά την άποψή μας συμπληρώνουν ε, ελλείψεις. Όμως, Στην έκθεσή μου δυστυχώς δεν κατάφερα να συμπεριλάβω όλες τις προτάσεις που έλαβα λόγω του περιορισμού που είχα. Η έκθεση αναφέρεται σε υψηλά επίπεδα φτώχεια, σε μεγάλο χάσμα ε, και τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε ανάγκη παρέμβασης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στην έκθεση αυτή Θέλουμε να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να επέλθει ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή. πρέπει ταυτόχρονα να γίνει ευκολότερη επιστροφή στην εργασία για εκείνους ε, οι οποίοι ήταν μακροχρόνια άνεργοι και επίσης να εξετάσουμε τις διαφορές ανάμεσα στη ζώνη του ευρώ και τις υπόλοιπες χώρες, να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να τα αναλύσουμε. Από την άλλη βέβαια χρειάζεται να τονιστεί ότι έχουν γίνει και βελτιώσεις και τις θετικές αυτές εξελίξεις πρέπει να τις ε, σχολιάσουμε αφού τις εντοπίσουμε και αυτές στην έκθεση. Πολλές προτάσεις και τροποποιήσεις κατέστησαν σαφές ε, πόσο διαφορετικές απόψεις έχουν οι διάφορες πολιτικές ομάδες. Οπότε θα ε, σταματήσω εδώ και θα δώσω το λόγο σε εσάς. Ο κύριος Χάρη Λόπες. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε για το ζήτημα αυτό εδώ στην Επιτροπή. Τώρα εδώ έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένε τροπολογίες. Εμείς θέλουμε απλώς να, θυμίσουμε ότι θα θέλαμε η έκθεση αυτή να αναφέρει ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε το έτος που μας μένει έτσι ώστε μια σειρά από ιδέες που έχουν συζητηθεί κατά τη διάρκεια θητείας να μπορέσουν να βρουν μια διέξοδο. Και η δυνατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να οδηγήσει σε συγκεκριμένες νομοθετικές ε, πράξεις, νομοθετικά μέτρα και δημοσιονομικά ε, για να επιλύσει μια σειρά από προβλήματα. Να πούμε επίσης ότι είναι αναγκαίο να καταπολεμήσουμε την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων, την ανισότητα γενικότερα ως ε, ένα στοιχείο ε, αποσταθεροποίησης ε, της οικονομίας μας και όλα αυτά να τα κάνουμε στα πλαίσια της έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ήθελα να προσθέσω ότι αυτό το εξάμεινο είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια που αρχίζουμε να διαπιστώνουμε κάποια ανησυχητικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τον οικονομικό κύκλο, ας πούμε, τις οικονομικές εξελίξεις. Πολλοί παράγοντες εξωτερικοί επέτρεψαν να έχουμε κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία τρία χρόνια αυτοί όμως οι παράγοντες ε, δεν ισχύουν πια. Οι τιμές ε, του πετρελαίου, η επεκτατική οικονομική πολιτική της ε, Κεντρικής Τράπεζας, τα χαμηλά επιτόκια, έχουν μια σειρά από στοιχεία που δείχνουν ότι οι δυνατότητες, η ρυθμοί ανάπτυξης, περιπτώσει χαλαρώνουν σχέση με τα τρία τελευταία χρόνια. Υπό αυτές λοιπόν τις προϋποθέσεις είναι πολύ σημαντικό, υπό αυτές τις συνθήκες, ε, να δώσουμε έμφαση στον, στην κοινωνική διάσταση που, έχουν, που έχει να κάνει με τις ε, πολιτικές, τις κοινωνικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα εργασιά, τις εργασιακές συνθήκες. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ η κυρία Μάκιντάι τώρα από, το, από την ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Σκιώδης ε, ε, η η συγκέντρια είναι η Αντρίκα του, του BCS, δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα όμω ε, και στη συγγνώμη γι' αυτό. Θα ήθελα όμω στο όνομά τη να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του και για το σχέδιο ε, των συμβασμών, συμβαστικών τροπολογιών που θα συζητηθεί αύριο το πρωί, αν κατάλαβα καλά, σε και των εισηγητών. Η ECR σε γενικέ γραμμέ υποστηρίζει την προσέγγιση τη εισηγήτρια και συμφωνεί και με το μεγαλύτερο μέρος των συμβαστικών κειμένων. Έχουμε όμως κάποιες ανησυχίες σε ό,τι αφορά τη διατύπωση ε, σε κάποιες παραγράφους, ιδιαίτερα ό,τι αφορά το συμβασμό 10 και το συμβασμό 11. Ε, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το θέμα της ευελιξίας, τη ρήτρα ευελιξίας και τη σχετική αναφορά στην ε, στο συμβασμό 12, όχι 11, 12. Για να χρησιμοποιηθεί αυτή η ρήτρα χρειάζονται πολύ, πολύ αυστηροί κανόνε. Κανένα από του τομεί μεταρρύθμιση που αναφέρονται ε, στο συμβαστικό κείμενο δεν πληρούν τι προποθέσει αυτέ. Παραδείγματο χάρη, η, λέμε ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να είναι μεγάλη, πρέπει να οδηγεί σε άμεση και μακροπρόθεσμη ε, αλλαγή δημοσιονομική. Ε, η ECR αντιμετωπίζει πρόβλημα και με τη διατύπωση στο 17, 19 και 20, σε αυτές τις προτάσεις συμβιβασμού. Πάντως ε, ο σκιός ηγητής θεωρεί ότι μπορούμε να, η σκιός για μας μπορεί, πιστεύει ότι μπορεί να βρεθεί συμβαστική λύση στην αυριανή συνάντηση, τελειώνοντας να πω ότι το ECR υποστηρίζει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της έκθεσης και ελπίζουμε να βρεθεί κοινό έδαφος για να υποστηρίξουμε και τον, την τελική μορφή που θα πάρει αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιο από του φιλελεύθερου. Ε, να πάμε απευθεία στους πράσινους. Η κυρία Λάμπερτ. Η κυρία Κούνεβα δεν είναι εδώ, έτσι. Ναι, η κυρία Λάμπερτ. Ναι, Πολλέ τροπολογίε είναι δική μας έμπνευση, ε, Πολλέ από αυτέ που ανέφερε η εισηγήτρια, αλλά και σε πέδο συμβαστικών κειμένων ε, ε, υπάρχει μια πολύ καλή βάση να βρεθεί δηλαδή συμβαστική λύση. Βεβαίω υπάρχει το θέμα του το γενικότερο ζήτημα των οικονομικών συνθήκων, αλλά υπάρχει και το θέμα του τι θα κάνουμε με τα χρήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή και πώ θα τα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να μειώσουμε τι ανισότητε. Αν οι ανισότητε ε, συνεχίσουν να αυξάνονται, τότε ε, δεν επιλύουμε και τίποτα. Δεν επιλύουμε κάποιο πρόβλημα στα πλαίσια του εξαμήνου. Εμεί λοιπόν επικεντρωθήκαμε ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή στι τροπολογίε μα ε, στο ζήτημα των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων, διότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν νωρί από την αγορά εργασία πριν από τη συνταξιδότησή του και αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τη διάκριση που υφίσταται λόγω τη ηλικία του και όχι λόγω επιλογή. Και βεβαίω ε, ε, συχνά αυτό οδηγεί και σε μη κατάλληλε συντάξει, μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, έκθεση σε φτώχεια και αυτό έχει να κάνει και ε, μια, ένα χάσμα ηλικιών που δημιουργείται. Ε, έχουμε ε, επίσης υποβάλει ένα από ό,τι αφορά την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες όπως αναφέρει η σύσταση για την ενεργή συμμετοχή όσων αποχωρούν από την αγορά εργασίας θα πρέπει και οι κυβερνήσεις μας να θυμηθούν κάποια πράγματα που είχαν πει ότι θα κάνουν το θέμα τώρα της πολιτικής συνοχής, ε, ε, το γεγονός ότι η οικονομική και η κοινωνική πολιτική πρέπει να πηγαίνει προς την κατεύθυνση και να ενισχυθεί το πυλώνος για τα κοινωνικά δικαιώματα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, καθώς και το θέμα της κοινωνία των πολιτών και τον διάλογο, του διαλόγου στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, από ό,τι φαίνεται, ε, δεν λαμβάνουν υπόψη επαρκώς ε, και θα πρέπει αυτό το λέει η έκθεση. Αναμένουμε τώρα τις ε, τροπολογίες. Ε, ελπίζω να βρεθούν ε, συμβαστικές λύσεις που θα βελτιώσουν το κείμενο. Ευχαριστώ. Να κλείσουμε τους και ε, Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να θέλει το λόγο. Ωραία. Αν δεν υπάρχει κανένας, να ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα να, να σας ευχαριστήσω όλους για τις παρατηρήσεις σας. Πραγματικά ήταν πολύ προσεκτικές αυτές οι παρατηρήσεις. Ιδιαίτερα τα σημεία αυτά που αφορούν κοινωνικά θέματα, κοινωνική ένταξη, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ένταξη όλων των κοινωνικών ομάδων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την ε, διαθεσιμότητά τους. Δίχως άλλο θα καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό τελικό κείμενο με πολύ καλές συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Μάλλον θα υιοθετηθεί στις 8 9 Οκτωβρίου και στην δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου θα γίνει η ψηφοφορία. Έχουμε 10 λεπτά διάλειμμα.

Okay.

Ευχαριστώ. Good afternoon again, colleagues. Καλησπέρα σας και πάλι αγαπητοί συνάδελφοι. Προτείνω να προχωρήσουμε στις σημερινές ψηφοφορίες. Η πρώτη αφορά την γνωμοδότηση για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση κάτω χώρες. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με 34 ψήφους υπέρ. Επόμενη ψηφοφορία για την έγκριση μιας επιστολής σχετικά με τις κοινέ διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και αρκετά άλλα ταμεία, καθώς επίσης και ορισμένες τροπολογίες. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω. Αποχές, με συγχωρείτε. Ας επαναλάβουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Μάλλον απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την επιστολή όπως έχει τροποποιηθεί. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά θέλετε. Πολύ ωραία. Καλύτερα ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνατε. Σας ευχαριστώ πολύ. περνάμε στο σχέδιο έκθεσης για το ρόλο της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επανένταξη των ανέργων. Συμβιβαστική τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές μάλλον εγκρίνεται θα ήθελα όμως να ελέγξουμε και ηλεκτρονικά Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Την 21 ψηφίζουμε. Υπέρ. Συμβιβαστική τροπολογία 21. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 85. Πέρας. Εγκρίνεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 95. Υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά πέρας απορρίπτεται Ninety 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά Yes, 98. Την 98 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Σαράντα εννιά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική δεκατέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική δεκαπέντε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Πέρασε και εγκρίνεται. Όλη, όλο το σχέδιο έκθεση. Όπω έχει τροποποιηθεί ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τώρα να περάσουμε την επόμενη ψηφοφορία το σχέδιο γνωμοδότησης για την προστασία των προσώπων ε, για, που, που αναφέρουν παραβίαση κοινοτικής νομοθεσίας. Δύο προφορικές τροπολογίες υπάρχουν. Θα τις αναφέρω όταν έρθει η ώρα τους. Συμβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαναλαμβάνουμε. Συμβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, τροπολογία 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβασμός 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 101. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο σκέλος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο σκέλος. Υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε αυτό, να το επαληθεύσουμε. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 καθώς και 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 15 υπέρ κατά αποχές να επαναλάβουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να το, να το επαληθεύσουμε αν θέλετε. Συμβιβασμός 15 λοιπόν. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία, εγκρίνεται. Συμβασμός 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να το παληθεύσουμε αυτό άρχιτη ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να το επαληθεύσουμε 124 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορία. εγκρίνεται 125 υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε και αυτό. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα στην 126 υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Θα την διαβάσω. Σε αυτές τις συναντήσεις ο αναφέρον θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνοδεύεται από έναν εκπρόσωπο της επιλογής του. Ο υπαλλήλος, ο εκπρόσωπος μάλλον του υπαλλήλου είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει τις πληροφορίες εμπιστευτικές και, και σε ασφάλεια. Έχει κάποιος ε, αντίρρηση? Ωραία, να ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 128 υπέρ κατά δεν είναι σαφές για μένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 9 υπέρ 10 εννοούσε η πρόεδρος, συμβιβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να το επαληθεύσουμε 132 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 133 σε δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, καλύτερα να το παληθεύσουμε και αυτό μετά τις αποχές, άρχη ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά καλύτερα να το παρθέσουμε άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται Εκατόν τριάντα πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται απορρίπτεται ναι αλλά ας το επαληθεύσουμε πέρας ψηφοφορίας όντως απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε παρακαλώ πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται συμβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ α όχι κατά πίπτη, συγγνώμη 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβασμός 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται αν θέλετε να το επαληθεύσουμε Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία και όντω απορρίπτεται. 190 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει και αυτό να το επαληθεύσουμε 190 λοιπόν άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας και όλους απορρίπτεται 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να το ελέγξουμε και αυτό άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 αποσύρθηκε 198 υπέρ κατά αποχές μάλλον εγκρίνεται ας το τσεκάρουμε όμως πέρας ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 200 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στο 201 τώρα έχουμε άλλη μια προφορική τροπολογία που αντικαθιστά τον όρο shall με may Δηλαδή δεν λέμε τα κράτη-μέλη θα εισαγάγουν, λέμε τα κράτη-μέλη μπορούν να εισαγάγουν. Και κάπου αλλού στο κείμενο δεν λέμε θα δημιουργήσει ένα σύστημα αναφορών, αλλά δύναται να δημιουργήσει. Να ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ναι, το 200 ήταν αυτό μαζί με την προφορική τροπολογία. Ναι, ναι, το 201 ήταν. Τώρα πάμε στο 202. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε καλύτερα το 31 ψηφίζουμε απορρίπτεται 18-23 32 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές υπέρ ξανά κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 σε δύο μέρη πρώτο σκέλος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά θα πρέπει να το επαληθεύσουμε το 50 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 σε 2 σκέλη το πρώτο σκέλος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο σκέλος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές για να το επαληθεύσουμε άχτη ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά η ίδια πλειοψηφία πρέπει να έχουμε εδώ αλλά στο το και ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 α είναι το ίδιο μάλιστα 61 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να το επαληθεύσουμε αυτό η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας και απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές και αυτό θα πρέπει να το επαληθεύσουμε άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με μία ψήφο 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται να το επαληθεύσουμε όμως η ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά εδώ επί του συνόλου. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται και έτσι Συνάδελφοι, ολοκληρώνει τη σημερινή συνεδρίαση. Ολοκληρώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.